il presidente sono pronte le schede allora επαναλαμβάνουμε τη σύνοδο ευχαριστώ έχουν τυπωθεί τα νέα ψηφοδελτία οπότε περνάμε στη δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή τριών αντιπροέδρων Πρέπει να αντικαταστήσουμε, να αντικαταστήσουμε την κυρία Τάλερ, μια ψηφολέκτρια που μα είπε ότι δυστυχώ ε, δεν μπορεί να έρθει, έχει ελμένε υποχρεώσει. Θα πρέπει λοιπόν να διορίσουμε τώρα ένα νέο ψηφολέκτη. Ονορεύολε Ρομπέρτα Μέτσολα. Η ε, κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα. Ε, Παρίσταται. Παρίσταται. Ονορεύολε Μέτσολα. Κυρία Μέτσολα. Δεν φαίνεται. Η κυρία Βάνα Πλούμπ. Okay. Το αποδέχεστε, αναλαμβάνετε την αρμοδιότητα. Ωραία λοιπόν, καλό τους ψηφολέκτες να λάβουν θέση δίπλα στις ε, κάλπες. Θα ψηφίσουν στο τέλος της ψηφοφορίας. Η κυρία Πλούμ, Ροβάνα Πλούμ, θα είναι στην κάλπη NR. Μπορεί να λάβει θέση. στη σχετική κάλπη δίπλα. Allora, ripetiamo eh, una, la regola. Επαναλαμβάνουμε τον κανόνα. Πρέπει να απονείμουμε τρεις θέσεις. Μπορείτε να ψηφίσετε τρεις υποψηφίους, το λιγότερο δύο. Ιδάλλως το ψηφοδέλτιο θα θεωρηθεί άκυρο. Να μοιραστούν τα ψηφοδέλτια, έχουν μοιραστεί μάλλον. AUTHORWAVE Allora la votazione è aperta. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται, άρχεται. Μπορείτε να ψηφίσετε.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 Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, οπότε αφού έληξε η ψηφοφορία, καλώ τους ψηφολέκτες να πάνε στην αίθουσα R01108 και διακόπτεται η σύνοδος.